Ο Πρόεδρος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, επαναλαμβάνεται η Σύνοδος. Τα χτεσινά πρακτικά και τα εγκεκριμένα κείμενα είναι διαθέσιμα. Εάν κανείς δεν θέλει να παρέμβει επ' αυτών, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά της χτεσινής ημέρας. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά μια κοινή συζήτηση για ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που μας απασχολούν